κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την εντολή του. Και εφόσον θα έχει δηλώσει γραπτό, ότι δεν έχει κάποιο αξίωμα ή ιδιότητα που να συγκρούεται με την ιδιότητά του ε, ως Ευρωβουλευτού και να καθιστά σύμβατη αυτή την ιδιότητα. Στις 20 ε, Φεβρουαρίου το ε, Κοινοβούλιο εξέτασε το, ε, την εντολή σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του συναδέλφου κυρίου Μάρκ Ντέμεσμέκερ και αυτό από την 1η Φεβρουαρίου 2013 επικυρώνει την εντολή. Προτείνω να επικυρωθεί αυτή η εντολή. Υπάρχουν ενστάσεις? Δεν υπάρχουν. Έτσι λοιπόν έχει κυρωθεί η εντολη υπαρχουν στασεις δεν υπαρχουν ετσι λοιπον εχει κυρωθει η εντολη η κυρία Μάρτα Αντρέασεν μου δήλωσε ότι από τις 25 Φεβρουαρίου δεν θα ανήκει πλέον στην Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας. Από τους σοσιαλδημοκράτες έχω ένα αίτημα η κυρία Φραντσέσκα Μπαρατσού να διοριστεί ως μέλος στην Επιτροπή.